ευχαριστούμε για την πρόταση και σας ευχαριστούμε κυρίως ε, για την υποστήριξή σας, τόσο ώστε να έχουμε τα, ενεργεια... τα ενεργειακά δίκτυα που χρειαζόμαστε για το 2020 και μετά. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε και ευχαριστώ και τον εισηγητή τον κύριο Σώσα Βάγκνερ και τώρα... Περνούμε στην επόμενη έκθεση που είναι η έκθεση του κυρίου Ντερόσα «Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος». Ε, παρακαλώ, θα θέλαμε να ακούσουμε τα εισαγωγικά σας σχόλια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους. Αυτή η έκθεση για το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος ε, μας προτείνει ρεαλιστικές ιδέες ε, για τις υπηρεσίες αυτές και για και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας ε, για τα άτομα που ασχολούνται σε αυτόν τον τομέα. Μιλάει για τους κοινωνικούς εταίρους, για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες, 285 τροπολογίες και ελπίζουμε να κρατήσουμε την ακαιρεότητα και την ουσία της έκθεσης ε, κατά την ψηφοφορία αύριο. Μπορεί να έχουμε διστάμενες απόψεις ε, και για νομικά θέματα και για θέματα αρχής, αλλά η ομάδα εργασία μας προτείνει μια μέθοδο ε, βιώσιμων λύσεων. Προτείνεται ένα φόρουμ για τις υπηρεσίες ε, γενικού συμφέροντος για να παρακολουθείτε η πρόοδο της ομάδας εργασίας και να υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό εθελοντικό πλαίσιο. Από την έρευνα αποδεικνύεται ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικότερα είναι ανεκτήμητες και έχουν και ζωτικό οικονομικό χαρακτήρα. Το 26% του ΑΕΠ αποτελούν και απασχολούν 64 εκατομμύρια άτομα, των οποίων το 1 τρίτο αποτελείται σε υπηρεσίε υγεία και κοινωνικού χαρακτήρα. Ο κοινωνικό τομέα ε, είναι πολύ σημαντικό γιατί διασφαλίζει την ένταξη στην κοινωνία και διευκολύνει την ε, συνοχή. Τονίζονται οι απαραίτητε ε, προσπάθειες για την εξέβρεση λύση. Υπάρχουν δυσκολίες από τους κανόνες για τις κρατικέ ενισχύσεις και για την διαδικασία δημοσίων συμβάσεων και στην έκθεση αναφέρονται οι ανεπάρκειες οι οποίες υπάρχουν. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, ε, διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων. Το 2007 ήταν η τελευταία φορά που αναφέρθηκε το θέμα των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος ε, στο ε, Κοινοβούλιο και στα τέλη του έτους κατέρευσε το, το πρόγραμμα το οποίο προωθούσε η Επιτροπή για το σύμβουλο τα τελευταία χρόνια και ήταν μεγάλο το οικονομικό κόστος. Μετά από την περίοδο εκείνη καταλήξαμε σε μια περίοδο κρίσης ε, με πολύ ε, δυσάρεστο χαρακτήρα. Υπάρχουν ε, πολλές πιέσεις για την χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών σε εποχές κρίσης και στην έκθεση αναφέρονται πιθανέ λύσεις. Λόγω της κρίσης και της έλλειψης απασχόλησης, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται περισσότερο από ποτέ την πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και χρειάζεται επίσης και η προστιθέμενη αξία την οποία μπορούν να μας δώσουν οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να προσαρμοστεί καταλήλως αυτή η έκθεση και περιμένω με ενδιαφέρον τη συνεργασία με όλους τους πολίτες ώστε να μπορέσουν να έχουν πραγματικά τις υπηρεσίες που τους ταιριάζουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κλείνοντας όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου, τους κοιόδης συζητητές και το προσωπικό, όλους εκείνους ε, τους εκπροσώπους τη κοινωνία των πολιτών που ε, συνεισέφεραν με χρήσιμε ιδέες και καινοτόμε ιδέε που ελπίζω ότι η ομάδα εργασία θα μπορέσει να διαμορφώσει κατά τον κατάλληλο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ντερόσα. Η κυρία Μπαστό έχει ζητήσει το λόγο. Είστε έτοιμοι να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση που συζητούμε τώρα έχει ιδιαίτερη σημασία λαμβάνοντα υπόψη την επιρροή που έχουν οι κοινωνικέ υπηρεσίε γενικού συμφέροντος στην καθημερινή ζωή των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και για την κοινωνική συνοχή, τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. Η συνεργασία με τον εισηγητή Πρόσια Δερόσα ήταν πραγματικά πάρα πολύ επικοδομητική και όπω είπε και ο ίδιο εισηγητή, διευκρίνησε πολλά σημεία και έτσι καταλήξαμε σε διάφορε συμβαστικέ λύσει στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων από το αποτέλεσμα που, των ε, διαπραγματεύσεων, δηλαδή την έκθεση, είμαστε ικανοποιημένοι και συγχαίρω τον εισηγητή. Η βασική μας ε, μέρημνα ήταν να διευκρινίσουμε ότι οι αρμοδιότητες σε αυτό το τομέα είναι εθνικές, οι εθνικές αρχές κατέχουν λοιπόν την ε, αρμοδιότητα της οργάνωσης και της χρηματοδότησης και του σχεδιασμού των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Ε, διείστανται οι απόψει ε, σε σχέση με την σκοπιμότητα του να έχουμε ευρωπαϊκέ κοινωνικέ υπηρεσίε ε, λόγω των εθνικών ιδιωτεροτήτων στον τομέα του, του τη υγεία, τη παιδεία, τη κοινωνική ασφάλιση. Πρέπει κάποιο να έχει βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρα. Είναι ο ακρογωνίο λήθο κάθε καλού σχεδιασμού τέτοια πολιτική. Σα ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εγκάρσια κοινωνική ρήτρα και το άρθρο 14 της Λισαβόνας δεσμευτικά εγγυώνται τα κοινωνικά δικαιώματα και τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Καιρός είναι λοιπόν να αποδείξουμε στους πολίτες ότι έχει ξεκινήσει η πορεία της κοινωνικής Ευρώπης γνωρίζοντας και τις ιδιαιτερότητες των κανόνων ανταγωνισμού. Αλλά να ξέρετε όμως όλες αυτές οι δραστηριότητες βασίζονται στην κοινωνία των πολιτών, είναι αρχές ριζωμένες Χρειάζεται λοιπόν παγκοσμιότητα, οικουμενικότητα και συλλογική δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες που αποτελούν παράγοντα ευημερία και κοινωνικής πρόοδου. Κυρία Επίτροπε, είπατε καιρός να μπούμε επί του συγκεκριμένου. Και συμφωνώ, προτείνω να έχουμε ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό σχέδιο για τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος σας καλώ λοιπόν να ψηφίσετε το, το εναλλακτικό ψήφισμα που κατέθεσε η ομάδα μου η πράσινη. Ε, ευχαριστώ. Κύριος Χάουιτ. Κύριε Πρόεδρε, σωστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να τονίσει το ρόλο του, τόσο ώστε να μην ε, φύγεται ο ανταγωνισμό και στο ψήφισμα αυτό θα πρέπει να προστατεύουμε θέματα που αφορούν και τη στέγαση και την υγεία. Χαιρετίζουμε τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην έκθεση και κάνουμε έκκληση να προστατεύσουμε τις, υπηρεσίες, τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας μας κατά των περικοπών σε αυτόν τον τομέα στις εποχές ε, δημοσιονομικής κρίσης. Ιδίως ε, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, θα χαρούν από μια τέτοια υποστήριξη εκ μέρους μας και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται αυτές οι υπηρεσίες και ξέρουμε ότι η ανάθεση και η ανάθεση συμβάσεων είναι ένας μόνο τρόπος για να παρασχεθούν αυτές ε, οι υπηρεσίες και δεν θα πρέπει μόνο το ελάχιστο δυνατό κόστος να είναι ε, ο γνώμων για την λήψη αποφάσεων Μέσω του ψηφίσματος αυτού μιλάμε για τα θέματα κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος ε, και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή και θα ήθελα κατά την ψηφοφορία να ληφθούν υπόψη όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Χαουίτη και κυρία Φιγκορέιντο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα αρχίστως να τονίσω την σημασία των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος ε, και γενικότερα των υπηρεσιών κοινή ωφελία. Ε, χωρίς αυτές δεν υπάρχει καμία ε, κοινωνική συνοχή, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα πρέπει να τροποποιήσουμε αυτές τις, πολιτικές, τις απελευθέρωση όλων των τομέων. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πολιτική κοινωνικής προόδου για να έχουμε ποιοτικέ καθολικές υπηρεσίες υπηρεσίες γενικού συμφέροντος ε, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία ε, στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση. Χρειαζόμαστε κατεπηγόντως μια αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων της απελευθέρωσης σε βασικούς τομείς επί της ζωής των πολιτών, ε, μεταφορές, ενέργεια, ε, υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική προστασία, όλοι αυτοί οι τομείς ε, και γι' αυτό περιμένουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις της Επιτρόπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είμαι σκιός συζητή από την Επιτροπή Ρέτζη και επι... Ε, χαιρετίζω την έκθεση του κυρίου Εντερόσα. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα βασικό πυλώνα της ε, ε, κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο αυτές οι υπηρεσίες για την κοινωνική συνοχή. Προφανέστατα δεν μπορούμε να έχουμε ελάχιστα επίπεδα προστασίας σε κάποια κράτη-μέλη και μόνο. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτό και πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται σεβαστές οι εθνικές, περιφερειακές και τομικές αρμοδιότητες στον τομέα των ε, καθολικών υπηρεσιών. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ε, ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και κάθε περιοχής για να καλύψει τις ανάγκες όλων των πολιτών. Ε, με σούσει της κρίσης προσπαθούν να φτιάξουν ένα δίχτυ ασφαλείας για τους λιγότερο ε, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι συγκεντρώνονται όλο ένα και περισσότερο οι εξουσίες, αποφασίζουν οι μεγάλοι οικονομικοί όμιλοι και δεν ε, ε, κατοχυρώνεται αυτή η δίκαιη πρόσβαση για όλους η Επίτροπος, ευχαριστώ. Παρακολούθησα ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση που έγινε στο Κοινοβούλιο για τι υπηρεσίε γενικού ενδιαφέροντο. και συμμεριζόμαστε απόλυτα την ε, άποψη του εισηγητή για τι υπηρεσίε αυτέ. Ε, συμφωνούμε ότι οι υπηρεσίες αυτές ε, παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην καθημερινή ζωή των πολιτών και έχουν κέριο ρόλο για να συμμετάσχουν όλοι στον καθημερινό βίο και να ασκούν τα βασικά του δικαιώματα. Συμφωνούμε με τον εισηγητή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να εγγυηθούμε ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικέ ε, ε, υπηρεσίε ε, για όλου, σε προσιτέ τιμέ. Ε, οπότε για τις γενικές υπηρεσίες ε, φυσικά θα υποπτεύουμε την εφαρμογή των ε, κείμενων διατάξεων αλλά επιπροσθέτως θεωρούμε με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να βοηθηθούν οι τους ώστε να οργανώσουν και να παράσχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες. Νομίζω ότι ότι υπάρχει και μεγάλη έλλειψη ενημέρωσης σε σχέση με την εφαρμογή των κανόνων και γι' αυτό τα τελευταία τέσσερα χρόνια φτιάξαμε νέα εργαλεία για να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση Προ προς όλους τους ενδιαφερομένους και θα συνεχίσουμε αυτέ τι προσπάθειε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση ε, ε, επανεξετάζει συγγνώμη, και αναθεωρεί τους κανόνες για τις κρατικές προμήθειες. Για τις κρατικές ε, προμήθειες θα μεριμνήσουμε ώστε να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες αυτό του τομέα του γενικού συμφέροντος και είναι σχετικά περιορισμένες οι στρεβλώσεις ανταγωνισμού σε αυτό το τομέα και αυτό θα ληφθεί υπόψη. Τον Μάρτιο ανακοινώσαμε τις ε, νέες ε, διατάξεις για ε, τις κρατικές προμήθειες και φυσικά προβλέπεται εξαίρεση για αυτές τις υπηρεσίες. Θέλουμε να διευκρινίσουμε λοιπόν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να μπορέσουμε να έχουμε ποιοτικές τέτοιες υπηρεσίες ε, και ελπίζω να σημειωθεί η πρόοδος ε, το ταχύτερο δυνατόν. Αναφερθήκατε στο φόρουμ για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και μιλήσατε για την ομάδα υψηλού επίπεδου που συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι μεταξύ των οποίων και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά όχι μόνο κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών από Επιτροπής. Πάντοτε είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για τους ε, κανόνες που θα διέπουν αυτές οι υπηρεσίες. Το δείξαμε εξάλλου στην ε, πρόσφατη διαβούλευση. Ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνεται σεβαστός ο ρόλος των οργάνων όπως προβλέπεται στη συνθήκη για να έχουμε και αυτά αποτελέσματα. Άρα κρίνουμε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό να ενισχύσουμε τις υφιστάμενες δομές και όχι να συγκροτήσουμε νέες, αλλά προτιθέμεθα να συζητήσουμε σε βάθος την μελλοντική οργάνωση των εργασιών μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Επίτροπε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ντερόσα, τον εισηγητή μας. Συνάδελφοι, έχω και καλά νέα. Ε, φτάσαμε στην τελευταία έκθεση για σήμερα. Ε, η έκθεση του κυρίου Κάτσμαδεκ, αντίκτυπος της αναπτυξιακής